έχετε παρατηρήσει όχι, θεωρούνται λοιπόν εγκεκριμένα. Έχω επίσης μια ανακοίνωση να σας κάνω. Έχω λάβει από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών διορισμό σε επιτροπή και